Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους βουλευτές εδώ. Θα ήθελα με την αδειά σας να περάσω στα αγγλικά, διότι καλός ή κακός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύουμε πολύ στα αγγλικά και πολλοί από τη δουλειά και τα έγγραφα που παράγουμε είναι στα αγγλικά. Είναι χαρά μου να σα παρουσιάσω σήμερα τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητα τη οδηγία πλαισίου για τα ύδατα, για το είδο. Ένα σημαντικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε 100.000 ε, αποθέματα επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό λεπτό να βρω το κουμπί μου και πώς να το κουνήσω. Εδώ λοιπόν αυτή η ευρεία ανάλυση δεν έχει να κάνει μόνο με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, που θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα και πλέον σφαιρικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό που ονομάζουμε και οι δύο οδηγίες ηθιγατρικές, δηλαδή αυτή για τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητα, ποιότητας, σημαντικά για να βλέπουμε και τη χημική σύσταση ε, των υδάτων και να μπορούμε να καταμετράμε την χημική ρήπανση και την οδηγία των υπογείων υδάτων, ε, πολύ σημαντική γιατί για το πόσιμο είδωρ τίνουμε να εξορίσουμε, να παίρνουμε το νερό από τους υδροφόρους ορίζοντες. Εδώ λοιπόν μας ενδιαφέρει η ποιοτική κατάσταση ε, των ε, υδάτων. Κοιτάζουμε να καλύψουμε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και επίσης ένα σημαντικό είναι πώς προχωρά και η οδηγία για τις πλημμύρες. Εδώ υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω των εξελίξεων που έρχονται από τις κλιματικές αλλαγές. Ταυτόχρονα θα διεξαγάγουμε και μία αξιολόγηση για την οδηγία της διαχείρισης αστικών λιμάτων. Μία οδηγία που είναι σημαντική και υποχρεώνει όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολούνται με την επεξεργασία των αστικών λιμάτων αλλά και κάποια βιομηχανικά λίματα. Ας κοιτάξουμε τώρα το πρώτο σκέλος, την ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Παραπάει γρήγορα. Ίσως δεν χρειάζεται να ακολουθώ τι διαφάνειε. Πρώτα απ' όλα, να πάω απευθεία στην επόμενη διαφάνεια. Να τονίσω ότι ω συνήθω σε όλη αυτή την προσπάθεια και με βάση τη αρχή τη καλύτερη νομοθεσία, έχουμε χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό διαθέσιμων πηγών πληροφοριών. Βλέπετε εδώ όλες αυτές τον κατάλογο. Θα ήθελα να τονίσω όμως την πολύ σημαντική έκθεση για την κατάσταση των υδάτων που δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος τον Ιούλιο του 2018. Η έκθεση αυτή ήρθε στην κατάλληλη χρονική στιγμή πριν την έκθεση του ΟΗΕ, την σημαντικότατη έκθεση του ΟΗΕ, για τους κινδύνους από την επίταση ε, των κλιματικών αλλαγών και την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Τα λάβαμε και τα δύο υπόψη, όπως και τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, που ε, διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν το 2018, μελέτες επίσης από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο. Ε, όλος αυτός ο έλεγχος καταλληλότητας είναι μία από τις μεγαλύτερες διαβουλεύσεις που διεξήγαμε το 2019 οδήγησαν σε 370.000 τουλάχιστον αποκρίσεις, τεράστιο δείγμα, που έχει να κάνει με την πολύ επιτυχημένη εκστρατεία ευαισθητοποίηση που, είχε ξεκινήσει, που είχαν ξεκινήσει περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και δείχνει βεβαίως και την ε, διάθεση να παραμείνει υψηλό το επίπεδο φιλοδοξία για αυτό το νομοθέτημα. Ήταν πολλέ οι συναντήσει βεβαίω και των ενδιαφερομένων, των εστιακών όπω ονομάζονται ομάδων και τουλάχιστον 100 έγγραφα θέσεων. Αυτή η διαδικασία διαβούλευση πραγματικά έλαβε πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον από του πολίτε του ίδιου. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποια από τα βασικά πορίσματα που αναλύσαμε στον έλεγχο καταλληλότητας. Αλλά πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι η καθοριστική το καθοριστικό επίτευγμα της οδηγίας αυτής από το 2000 είναι ότι κατάφερε να επιτρέψει τη δημιουργία ανά την Ευρώπη διαρθρώσεων δομών διαχείρισης για την κοινή ακριβώς διαχείριση των λεκανών ποταμών για τις κήτες των ποταμών. Εδώ καταφέραμε 60% αυτών των λεκανών και των κοιτών να να τα διαχειριζόμαστε από κοινού, γιατί βρίσκονται σε, στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών τι περισσότερες φορές. Είναι σημαντικό λοιπόν τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται αποτελεσματικά και επιτυχώς, προκειμένου να διαχειρίζονται σωστά τα ύδατα. Ωστόσο, το λιγότερο ενθαρρυντικό είναι ότι η υλοποίηση αυτή τη οδηγία δεν ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο ελπίσαμε. Το 2000 είχαν ε, υποσχεθεί τα κράτη-μέλη να ε, πετύχουν καλό επίπεδο για όλη τη διαχείριση των υδατινών πόρων στο 2015. Δεν έχουμε φτάσει όμως ακόμα εκεί. Νομικώς έχουν τη δυνατότητα βάσει του άρθρου 4 της ε, οδηγίας αυτής να πετύχουν την καλή κατάσταση που θέλαμε. Ως το 2027 έχουν αυτό το περιθώριο. Όμως υπάρχουν δομικά προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το σύνολο, το ποσό χρηματοδότησης που διαθέτουν για να λάβουν κάποια μέτρα που απαιτούνται, όπως την αποκατάσταση των φυσικών πόρων ή την αντιμετώπιση κάποιων ε, πιέσεων σε επίπεδο γεωμορφολογικό και επίσης κάτι άλλο που εντοπίσαμε στον έλεγχο καταλληλότητας, ότι οι στόχοι για τα ύβατα δεν έχουν ενταχθεί επαρκώς σε άλλες διευθυντικές πολιτικές πολιτικές επίσης σημαντικές, όπως αυτές που εντοπίσαμε στο κεφάλαιο της συνοχής. Δηλαδή, οι στόχοι για το νερό θα μπορούσαν να συνδυαστούν με την ενεργειακή, τη γεωργική πολιτική και ακόμη με την πολιτική μεταφορών. Τώρα, η οδηγία για τις πλημμύρες. Από τον έλεγχο καταλήξαμε ότι αφού η οδηγία έχει περάσει μόνο στον πρώτο της κύκλο υλοποίηση, ε, παρά είναι νωρί για να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα για το κατά πόσον είναι κατάλληλη και σκόπιμη, ε, όπως αρχικά σχεδιάστηκε, αλλά δεν είναι και πολύ αργά για να δούμε κατά πόσον είχε έναν θετικό ε, αντίκτυπο στο πώς τα κράτη-μέλη χαράσουν και ε, εκπονούν τα ε, προγράμματα αντιμετώπισης των πλημμυρών. Ιδίω εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος ή απειλή από πλημμύρες. Ταυτόχρονα η απειλη απο πλημμυρε ταυτοχρονα Επιτροπή το 2018 φρόντισε να κάνει διεξοδική ανάλυση όλων των δευτερογενών προγραμμάτων διαχείρισης και ποταμών, ώστε αυτά που εμπίπταν στον, στην οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων και στα πρώτα σχέδια διαχείριση. Έχει μάλιστα εκδώσει συστάσεις προ τα κάτι μέλη και σε ό,τι αφορά τι πλημμύρε, βλέπουμε ότι μόνο μια μικρή, ένα μικρό ποσοστό κρατών μελών είναι σήμερα σε θέση να ε, συνδυάσουν τα πρότυπα που έχουν προκύψει από τις ανάγκες αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών με την αντιμετώπιση των πλημμυρών και τα προγράμματά τους. Προσπαθήσαμε εδώ όλα να τα ανακεφαλαιώσουμε σε στήλε, για να το πω έτσι, σε τομεί όπου έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχο καταλληλότητα και να δούμε τι πορίσματα μπορούμε να αντλήσουμε. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι η οδηγία έχει επιφέρει θετικά βήματα πρόοδου, αλλά πιο ε, αργά, βραδέως, σε σχέση με αυτό που αρχικά επιθύμησαν οι νομοθέτες. Η οδηγία Ε, αυτή συμπεριέχει την ε, one in all out ε, αρχή, δηλαδή αν μία από τις παραμέτρους την οποία ελέγχουμε σε σχέση με τα ύδατα δεν ακολουθείται, δεν τηρείται πλήρως, τότε δεν μπορούμε να, να πούμε ότι μια λεκάνη, μια κήτη είναι πλήρως σε καλή κατάσταση, όμως πρέπει να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Έχουμε δει σωματικές Μειώσει ε, στην παρουσία βαρέων μετάλλων σε κάποιες περιπτώσεις υδατινών πόρων ή κάποιων σοβαρών ρήπων όπως του υδρακύρου ε, που παραμένει Εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι η χημική κατάσταση, η χημική υγεία είναι απόλυτα καλή, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξουμε το χρόνο. Επίση, η οδηγία δίνει μεν κάποιε γενικά συντευτήριε γραμμέ, είναι όμω και διαλεκτική ευέλικτη. Δηλαδή, θέλουμε στενότερες σχέσεις συνεργασίας ε, και βλέπουμε να υπάρχει περιθώριο ε, περαιτέρω αναπτυξή του. Όμω είναι σαφέ ότι τα προγράμματα διαχείριση των κοιτών των ποταμών ε, έχουν ε, πονηθεί έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν περιθώριο να εντάξουν εκεί και τι διάφορε μέρημνε περί κλιματικών αλλαγών που έχουν ανακύψει. Και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό επίπεδο. Επίση, έχουμε εντοπίσει κάποιε αναδυόμενε μέρημνε, τι οποίε έχουμε ονομάσει, αναδυόμενου νέου ρήπου, δηλαδή από ουσίε φαρμακολογικές ή μικροπλαστικά και είμαστε σε μια φάση καλή για την υλοποίηση της οδηγίας αυτής. Γιατί την η τελευταία προθεσμία ώστε τα κράτη-μέλη να πετύχουν την πλήρη συμμόρφωση το 2027. Οπότε, στη φάση αυτή τα κράτη-μέλη είναι τουλάχιστον στη φάση εκπόνηση των του τρίτου κύκλου προγραμμάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων και σημειώνουμε ότι υπάρχει μια ευρύτατη ε, αξιοποίηση της δυνατότητας να ε, χρησιμοποιηθεί η αρχή να αξιοποιηθούν οι εξαιρέσει που προσφέρει η οδηγία αυτή, ώστε να κηρυχθεί η κατάσταση κάποιων κοιτών ποταμών καλή για κάποιον αριθμό ετών. 50% τουλάχιστον αυτή τη στιγμή των υδάτινων πόρων μα υποφελούνται από αυτή την εξαίρεση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη υλοποίηση, καλύτερη κοινή εφαρμογή τη οδηγία σε όλα τα κατημέλη, μελη σε συνεργασία μεταξύ του. Υπάρχουν βελτιώσει στο επίπεδο των χημικών ουσιών. Είδαμε με τον έλεγχο καταλληλότητα λόγου χάρη ότι τα πρότυπα περιβαλλοντική ποιότητα που, έχει έχουν δημιουργήσει έναν πολύ καλό κατάλογο ε, παρακολούθησης κάποιων συγκεκριμένων τοξικών ουσιών και της παρουσίας τους σε υδατινούς πόρους, δεν μας επέτρεπε να δούμε αρκετά το κατά πόσον η ανάμιξη, ο συνδυασμός κάποιων χημικών ουσιών μπορεί να είναι μια απειλή αυτό μα απασχολεί τώρα ή επίση οποιαδήποτε επικαιροποίηση των παραρτημάτων αυτής της τη θηγατρική εντό εισαγωγικών οδηγία που επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των χημικών ουσιών και τη παρουσία τους. Αυτά απαιτούν μια μακροσκελή και χρονοβόρα νομοθετική διαδικασία, οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όσο, το όσο γρήγορα θα θέλαμε. Και επίσης πρέπει οι στόχοι να συνδυαστούν ε, και στις διασυνοριακέ υδάτινε μεταφορέ, στην πολιτική μεταφορά, στην περιβαλλοντική πολιτική. Σκεφτείτε την εσωτερική ναυσιπλοεία λόγου χάρη πόσο σημαντική είναι και γι' αυτό θέλουμε να στραφούμε σε όλους ε, που συμμετέχουν και να τους θυμίσουμε το άρθρο 9 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ήδατα, που επί της αρχής προβλέπει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, υπολογίζουν την διασταυρούμενη ανάκτηση ε, δυνατοτήτων χρήσης των υδατινών πόρων λόγω της χρήσης στη γεωργία ή από τα νοικοκυριά. Εκεί λοιπόν στην Ευρώπη παραμένει λιγότερη δυνατότητα, παραμένουν λιγότερα περιθώρια για να επιταχύνουν την δράση τους και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε όμως τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Υπάρχουν και άλλα μέσα πλέον σήμερα, τεχνητή ε, ευθεία, η εξόριξη δεδομένων και πολλά άλλα που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη δουλειά των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. So I will... Ωραία λοιπόν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Έχω στον κατάλογο μου τον Κρίστοφ Χένσεν από το ΕΛΚ. Από τους σοσιαλιστές κανείς. Η Ρίκα Μίλλερ από τη Renew. Ο κύριος Γκίγκολτ από τους Πράσινους. και από την ΚΟΕ. Η Μα... Ποιος? Η Μαντλέν? Ο Μάλιν Μπιόρκ, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Μανφρέντι για την εξαιρετικά λεπτομερή παρουσίαση που έκανε. Η πόροι υδάτινοι της Ευρώπης ε, αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της αλλαγής του κλίματος, της αύξησης του πληθυσμού, της ε, αστικοποίησης, όπως επίσης και της αλλαγής των ε, οικονομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν τα τρίτα σχέδια για τη διαχείριση των ποταμών και Νομίζω πως θα κατατεθούν μέχρι τα τέλη του 2021, όπως είπε και η κυρία Μανφρέντη. Πείτε μου λοιπόν, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να έχουμε νομική βεβαιότητα, έτσι ώστε τα σχέδια αυτά να είναι παρκώς φιλόδοξα και να προφτάσουμε την προθεσμία του 20.000, του 2027. Και δεύτερη ερώτηση. Οι ενδιαφερόμενοι και οι επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει το επίπεδο φιλοδοξίας ε, και να μην ξανανοίξει την οδηγία ε, για τα ύδατα, γιατί φοβούνται πως τα κράτη-μέλη μπορεί να μειώσουν το επίπεδο φιλοδοξίας ε, σε σχέση με το παρελθόν. Και δεδομένου του Green Deal, θα ήθελα να μου πείτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επιθυμεί να ξανανοίξει αυτή την οδογία και αν την ανοίξει, ε, τι χρονοδιάγραμμα έχετε κατά νου. Από τη Ρινιού, Ενρίκα Μίλλερ. Ευχαριστούμε κυρία Μανφρέντι ο έλεγχος καταλληλότητας για την, της οδηγίας δείχνει ότι η επίτευξη των στόχων δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και δεν έχουν ενσωματωθεί σε άλλες ε, πολιτικές. Συγκεκριμένα αναφέρατε τη γεωργική πολιτική Και εκεί για το συνδυασμό με την γεωργική πολιτική έχει κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες καινούργιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να προστατεύουμε καλύτερα ε, με δείκτες τους υδάτινους πόρους. Θεωρείτε ότι όσα έχουν γίνει ως τώρα είναι αρκετά ή όχι και μήπως θα έπρεπε να ασκήσουμε περισσότερη πίεση για την ε, όλη διαδικασία εφόσον τώρα έχουμε και την αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής. Θα επιβαρυνθεί αυτή η αναθεώρηση ή όχι. Και μήπως χρειάζονται οδηγίες ε, που να επικεντρώνται σε τοπικότερο επίπεδο. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε μήπως το μέλλον της αγροτικής πολιτικής μπορεί από αυτά που αναφέρατε κι εσείς να επηρεαστεί, την παρουσία χημικών ουσιών από φαρμακολογικές πηγές, ή μικροπλαστικά, και να δούμε επίσης πόσο θα περιορίσουμε και το κόστος της διαχείρισης των υδάτων. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Τι δυνατότητες λοιπόν διαβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, ώστε στο μέλλον ιδίω οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις να υποστηρίξουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Πράσινη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, τόσο λεπτομερή απάντηση, λέει η κυρία Άουκεν, γιατί είναι εξαιρετική η οδηγία αυτή και είναι πολύ σημαντικό να μην αποδυναμωθεί, γιατί έχει αναβληθεί αρκετές φορές επειδή δεν είχαμε επαρκές επίπεδο εφαρμογής και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπερβολικά ευγενική με τα κράτη-μέλη και δέχτηκε τις διάφορες ε, προφάσεις που προβάλλουν. Στη Δανία λένε πως είναι η Γεωργία, όπου βρίσκουν με ιδιαίτερα πολυμήχανο τρόπο και καινούριου ε, λόγους για να μην εφαρμόσουν την οδηγία αυτή. Ελπίζω πως σύντομα πάντως θα πιέσετε έτσι ώστε να σεβαστούμε και τις προθεσμίες του 2027 και να μην δεχτείτε άλλες ε, αναβολές. Νομίζω ότι η παρουσίαση σας μας έδωσε ε, κάποια χέγγια έτσι ώστε να μην ξανανοίξει το κομμάτι αυτό, να μην κερδίσουν στο σημείο αυτό τα λόμπι, αλλά δεν βρήκα τα χημικά ε, κάπου σε αυτά που συζητήσατε. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ανοίξουμε την οδηγία. Αν τις τοποθετήσουμε στις ομάδες ουσιών και όχι μία-μία, θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Και μία τελευταία ερώτηση. Σας παρακαλώ, μην την ξανανοίξετε την οδηγία και να είστε και ε, σκληρή με τα κράτη-μέλη αν προσπαθήσουν να την αποφύγουν. Από το 2015 και μετά έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Οπότε πραγματικά η κατάσταση δεν είναι θετική. Και αν ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος εφαρμογής, όσο καθυστερούμε τόσο πιο πολύ αυξάνεται το κόστος αυτό. Και είναι και μεγαλύτερα τα επίπεδα ρήπανσης τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Ε, Μαλέν Μπιόρκ για την ΚΟΕ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Η οδηγία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, το λένε και οι υπεύθυνοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν τεράστια η, τεράστιο το ενδιαφέρον που έδειξαν οι πολίτες. Ε, ε, θέλησαν να εκφράσουν μαζικά τη γνώμη τους και είδατε, <laughs> μιλάω σου ειδικά, το λέω αυτό γιατί οι πολίτες μας ενδιαφέρονται και νομίζω ότι έλαβαν και μια σαφή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά όπως και προλαλή προλαλήσασα πότε θα πείτε απερίφραστα πως δεν θα ξανανοίξετε την οδηγία. Δεν περιμένουν την απάντηση αυτή μόνο οι πολίτες. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να αλλάξουν ε, σχέδια και να λάβουν ένα ε, περίφραστο μήνυμα για να δούμε τι θα γίνει με τους στόχους και πώς μπορούμε να αποφύγουμε ακόμα περισσότερες αναβολές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2027 για να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή. Και όπως μας δείξατε κι εσείς με την παρουσίαση που κάνετε, η στήριξη είναι μεγάλη και δεν φταίει το νομικό κείμενο για οποιαδήποτε προβλήματα με την εφαρμογή. Είναι μια σειρά άλλων θεμάτων που έχει προκύψει. Επαναλαμβάνω λοιπόν πως κατανοώ πως υπάρχει μεγάλη πίεση από τη βιομηχανία, από τα λόμπι, από τους γεωργούς και από αλλού. Και όλοι προσπαθούν να χαλα... Ε, ρώσουν ε, τις διατάξεις της οδηγίας αυτής, αλλά το μήνυμα που έχουμε λάβει από τους πολίτες είναι το εξής. Θέλουν να εφαρμοστεί. Μας ρωτάνε πού θα εστιάσει και δεν θέλει να συνεχίσουμε με business as usual. Πρέπει να καταλάβουν ότι το Green Deal κάτι σημαίνει, πώς θα εφαρμοστεί και είπαμε όχι νέα νομοθεσία, ναι στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε, έτσι ώστε η οδηγία αυτή να τηρηθεί. Το 50% της οδηγίας είναι εξαιρέσεις και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια και για όσους μας ακούνε σήμερα αυτό ζητάνε και εκείνοι. Μεγαλύτερη σαφήνεια.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 Στην, Ελλάδα, στην Ευρώπη συγγνώμη, έχουμε ένα σωρό κανόνε ε, για την προστασία του περιβάλλοντο, για την προστασία των υδάτινων πόρων. Και όμω ο έλεγχο καταλληλότητα ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι τουλάχιστον ε, μισέ των υδάτινων επιφανειών τη Ένωση δεν είναι σε καλή κατάσταση. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση για μία μόνο πτυχή των, υδάτικο, των υδάτινων πόρων ξεκίνησε διαδικασία που παραβάσει κατά τη Γερμανία. Ταυτόχρονα είναι τρομακτικό ότι 20 χρόνια μετά την ε, έγκριση και την θέση σε ισχύ αυτών των κανόνων δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες αυτές. Η καλή οικολογική κατάσταση έπρεπε να έχει επιτευχθεί το 2015 και τελικά υπάρχουν διαρκώς εξαιρέσεις και παρατάσεις. Στην δική σας ανάλυση ως τώρα μας λείπει η ανάλυση της μεθοδολογίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί ως τώρα δεν υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάση κατά των άλλων κρατών μελών όπου βλέπουμε ότι εμφανώς δεν έχουν, σεβαστεί και επιτευχθεί, δεν έχουν γίνει σεβαστοί και επιτευχθεί στόχοι. Γιατί ειδικά ε, μόνο στη Γερμανία, γιατί είναι ε, σαφές ότι ούτε το 2027 θα έχουν ε, φτάσει να σέβονται τους κανόνες. Στην δική μου την εκλογική ε, περιφέρεια υπήρξαν τουλάχιστον εκατοντάδε διαδικασίε παραβάση και όμως πού είναι οι ε, Πού είναι οι σοβαρέ συνέπειε. Εμένα λοιπόν η ερώτησή μου είναι θα αλλάξετε τη μεθοδολογία σα, τον τρόπο που εργάζεστε για να γίνει κάτι για αυτή την οδηγία πλαίσιο των ε, υδάτων και να επιβάλλονται κυρώσει, να είναι πιο ταχύε οι διαδικασίε. Διότι χωρί κυρώσει, ε, το 2027 πάλι εδώ θα καθόμαστε και θα λέμε τα ίδια. Άρα, ε, πώ αξιολογείτε την ίδια σα την μεθοδολογία, τον τρόπο που εργάζεστε εσεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα κάνετε για να επιταχύνετε και να κάνετε πιο ε, αποτελεσματικέ τι διαδικασίε παραβάση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστούμε για τους πρασίνους, η κυρία Παύλους. Ναι, και εδώ είδαμε ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την καταλληλότητα. όμως όταν έχουμε νόμος πρέπει να κοιτάζουμε ακριβώς και την εφαρμογή τους. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, ε, ο οργανισμός περιβάλλοντος ε, είχε εντοπίσει ότι είναι σημαντική λειτουργία των ποταμών για την παρουσία των υδάτινων οργανισμών επίσης και του φυτοπλανκτών και ότι πρέπει να προβλέψει κανείς τρόπους ενίσχυσης της προστασίας των υδάτινων πόρων όταν οι δευτερογενεί λειτουργίε των υδάτινων πόρων δεν λαμβάνονται επαρκώ υπόψη, χάνουμε μεγάλε δυνατότητε εξοικονόμηση πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν, επειδή η έκθεση του Οργανισμού Περιβάλλοντος το έδειξε και το είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας, υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν σχέση με τις χημικές ουσίες που καταλήγουν στους υδάτινους πόρους, που δεν αντιμετωπίζουν ε, ως προτεραιότητα τα κράτη-μέλη και επίσης πολύ μεγάλη είναι η μόλυνση από τα φαρμακευτικά προϊόντα που καταλήγουν στο νερό, κάτι που έχει ξεκινήσει να μελετάται από την δεκαετία του 80. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι για την αντιμετώπιση αυτών των χημικών όπως των πολυχλωρικών και για τις ουσίες που έχουν μεγάλη παρουσία στις κοίτες των ποταμών και τα εδάφη του περιβάλλοντος και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστούν από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν. Τα μικροπλαστικά καταλήγουν, όπως ξέρουμε, στα ψάρια και σε άλλους εδάφινους οργανισμούς. Τι έχετε σκοπό να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μανφρέντη για την παρουσίασή τη. Και πραγματικά ανησυχώ, ανησυχώ πάρα πολύ που διαβάζω ότι το σύνολο των κρατών μελών σήμερα έχουν ζητήσει ουσιαστικά παράταση. Παράταση για να επιτύχουν του στόχου του και να έχουν καλή κατάσταση και ποιότητα στα επιφανειακά ύδατα κυρίω. Με ανησυχεί ότι κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη είχαν κατά 90% ε, ζητήσει τα υδάτινα σώματα της επιφανείας να ε, συμπεριληφθούν στον πρώτο γύρο, στην πρώτη φάση επίτευξη των στόχων. Φαίνεται λοιπόν ότι για το νερό των ποταμών και λιμνών, το γλυκό νερό, έχουμε 4% ε, μείωση κατά ε, έτος, το μισό τουλάχιστον από ό,τι συμβαίνει με τα θαλάσσια ύδατα και ένα από τα τρία είδη που ζουν στο γλυκό νερό, τα τρία είδη ψαριών, απειλούνται με εξαφάνιση. Εδώ λοιπόν ξέρω την περίπτωση 370.000 πολιτών από τη δική μου περιφέρεια που ζητούν την προστασία των ποταμών, των λιμνών, των υδάτων μας και την προστασία της βιοποικιλότητάς μας. Ε, είναι σημαντική η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δει αν όντως λειτουργεί καλά η ισχύουσα οδηγία και πώ πρέπει να προχωρήσουμε με την εφαρμογή τη. Πρέπει να κάνουμε παραπάνω όμω. Κανένα βήμα οπισθοχώρηση, κανένα καμία ε, απόπειρα αποδυνάμωσης της οδηγίας δεν πρέπει να αποδεχθούμε σε σχέση με το πόσο ήδη είναι ευέλικτη και διαλλακτική. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε είναι οι δράσει προτεραιότητα που έχετε προβλέψει για να ενισχύσετε τα κράτη-μέλη και να υπάρξει μια σωστή ε, εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ποιότητα των υδάτων. Και πώ θα το πετύχετε, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να επικαιροποιήσετε την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Εκεί θα μπορούσαμε να πετύχουμε μείωση και ε, της παρουσίας των ε, ουσιών από φάρμακα και των μικροπλαστικών στα νερά, στα ύδατα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας. Έχετε ένα τέταρτο στη διάθεσή σας και θα γίνει και η συζήτηση για τα αστικά απόβλητα. Δεν ξέρω αν λίματα με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να απαντήσετε. Ε, αυτό το κάνω για να μπορέσουμε να κλείσουμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή, ε, να μιλήσω και για τα λύματα, γιατί ε, κάποιες ερωτήσεις έχουν πιο πολύ να κάνουν με τα λύματα. Λοιπόν, μιλώ τώρα αγγλικά και λέω πώς θα τα πω θεματικά. Καταρχήν, η βασική ερώτηση από εσά είναι εάν θα πούμε απερίφραστα πως δεν θα ξανανοίξουμε αυτή την οδηγία. Να σας πω λοιπόν το εξής. Ο έλεγχος καταλληλότητας καταλήγει πως η οδηγία για τα ύδατα είναι κατάλληλη, αλλά έχουμε εντοπίσει κάποια σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Και είναι δίκαιο να σας πω πως αυτή τη στιγμή συζητάμε με την πολιτική μας ηγησία τα θέματα αυτά όχι για να ρισκάρουμε να νερώσουμε την οδηγία αυτή, αλλά για να αξιολογήσουμε όλες τις εναλλακτικέ δυνατότητες που έχουμε στα πλαίσια του Green Deal που θα επικυρωθεί την ημέρα μετά τη δημοσίευση ε, των όσων θα κάνουμε την οδηγία αυτή. Έτσι ώστε το εργαλείο τούτο να μας επιτρέψει να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα και τους ε, κλιματικούς στόχους και τη βιοπικιλότητα που επιδιώκουμε όλοι για την Ευρώπη. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ευρύτερη συζήτηση που γίνεται με όλους σας και χαίρομαι πολύ που ακούω όλες τις απόψεις σας, τρέχουν συζητήσεις και με το Συμβούλιο, ίσως ξέρετε πως το Συμβούλιο σχεδιάζει να κάνει μία συζήτηση προς ανατολισμού στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος το Μάρτιο, συζητάμε αυτή τη στιγμή όλες τις απόψεις που έχουν συγκεντρωθεί τώρα που δημοσιεύσαμε τον έλεγχο καταλληλότητας έτσι ώστε να ακολουθήσουμε την άγουσα που θα μας δείξουν και να μας υποδείξουν στα πλαίσια του Green Deal. Τώρα, επιβολή παραβιάσεις. Έχουμε καταλήξει με το fitness check πως σε εθνική εφαρμογή μπορούν να γίνουν πολλά σε αυτό το επίπεδο. Και έχουμε ζητήσει στα πλαίσια του ερωτηματολογίου για τους ε, ενδιαφερόμενους τι πιστεύουν. Ποιο θα πρέπει να είναι το επίπεδο των κυρώσεων που δυνητικά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και από τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που έχουμε παραβιάσεις και η απάντηση είναι πως πολλοί πιστεύουν πως δεν είναι αρκετά αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές. Δεν ξέρω αν αυτό ταυτίζεται με τα παραδείγματα που δώσατε εσείς με άσχημες ιστορίες που έχουν διαπιστώσει με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Πολλές περιπτώσεις, κάποιες φορές και πολύ καθυστερημένα φτάνουν και στα αυτιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας εγγυηθώ πως είμαστε αποφασιστικοί, θα διώκουμε τις περιπτώσεις παραβίασης. Έχουμε αρκετές υποθέσεις που τρέχουν και το Φεβρουάριο του 19 εγκρίναμε μία σύσταση πολύ αυστηρή προς όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να τις καθοδηγήσουμε, να καθοδηγήσουμε τις αρχές τώρα που προετοιμάζουν αυτά τα σχέδια και σε εσωτερικό επίπεδο παρακολουθούμε στενά όλες τις ελλείψεις που έχουμε διαπιστώσει στα δεύτερα διαχειριστικά σχέδια για τα ε, για τους ποταμούς και πρέπει να σας πω πως η πολιτική μας για τις παραβιάσεις μας υποχρεώνει σε περίπτωση που υπάρχει διαστρωτική αποτυχία από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούμε το εργαλείο τούτο. Αλλά η πρωταρχική ευθύνη βαρύνει τα κράτη-μέλη. Επίσης, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει παντού το ίδιο επίπεδο δυναμισμού από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ έτσι ώστε να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την οδηγία αυτή στην πρακτική εφαρμογή. Τα έχουμε όλα κατά νου, τα συζητάμε και σε οριζόντιο επίπεδο γιατί είναι θέματα που αφορούν και άλλα τμήματα του περιβαλλοντικού στην αξιότιμη κυρία Μίλλερ θα απαντήσω πως η πρότασή μας για την ΚΑΠ και ο συσχετισμός με τις προτάσεις εδώ έχουν δημιουργήσει σύνδεσμο ερησιμότητας για την ε, χορήγηση παραπάνω κονδυλίων και επιδοτήσεων στους γεωργούς σε περίπτωση που σέβονται κάποια επιπλέον κριτήρια φιλικά προς το περιβάλλον. Θα σας αφήσω βέβαια, είστε συνομοθέτες, οι πολύ δραστήριοι στο φάκελο αυτό. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σας άκουσα, άκουσα πάρα πολλά σχόλια επίσης για τα χημικά, για τη χημική ρήπανση. Όντως αλλά στον έλεγχο καταλληλότητας το έχουμε εντοπίσει αυτό και έχουμε πει εδώ θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα σε συλλογικό επίπεδο και να αξιολογήσουμε ε, το σύνολο του αποτελέσματο που έχουν το μείγμα ουσιών στο νερό. Έχουμε ένα περιθώριο ελιγμών εκεί, αλλά θέλουμε να, ε, ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα στην πηγή. Ενδοκρινικοί διαταράκτες. Εδώ οι δύο συνάδελφοι με τους οποίους κάνουμε πολύ ε, ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για το πόσιμο νερό ξέρουν πως τα PCP και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες προσπαθούμε να του αντιμετωπίσουμε με μια ολιστική προσέγγιση και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το όσο έχει κάνει και για την ε, ε, ένδυα ύδατος στην οδηγία αυτή έχουμε και ποσοτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να σεβόμαστε και αυτά σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που κάνουμε για να σχεδιάσουμε την επόμενη στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπου θα αντιμετωπίσουμε ε, και το θέμα της ε, ένδυας υδάτων. Να σας προτείνω κυρία Πρόεδρε να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις με συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί και για την αξιολόγηση εγώ δεν έλαβα κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ <laughs> έχω να κάνω μια σχετική ερώτηση.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 Ευχαριστούμε. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη συζήτηση και να περάσουμε στον προπολογισμό του 2021 σε δύο λεφτά.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 Να σας πω λοιπόν πως θα μπορούσαμε να έχουμε στην κυροσύνη ένα φόρο. Είναι κάτι το οποίο ε, είχε αναφερθεί και ως ε, ε, φόρος επί των πιστωτικών υπηρεσιών ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, φόρο για τον διοξείδιο του άνθρακα στα σύνορα, ε, φόρο για το πλαστικό. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Είναι θέματα τα οποία επεξεργάζεται η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα έδιναν κέρδη στην Ευρώπη. Η Επιτροπή μας καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα κέρδη Ε, των εταιριών έχουν αυξηθεί ε, αλματοδός τα τελευταία χρόνια και παρόλα αυτά δεν μοιράζονται στους εργαζομένους, δεν επανεπενδύονται. Ε, λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει χρήμα για το κλίμα και παρόλα αυτά βλέπετε πως τα μερίσματα αυξάνονται και τα κέρδη δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλά. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί και ο Ρούσβελτ όταν ανέλαβε την εξουσία έριξαν όλοι τους φόρους. Δηλαδή η Φλόριντα και όλοι, οι, όλοι τα, όλες οι υπόλοιπες πολιτείες. Και τότε είπε μετά από τέσσερα χρόνια ο Ρούσβελτ ότι Φλόριντα, Τέξας, ομόσπονδος ε, φόρος 38%. Το είχε πει και ο Επίτροπος Μόντι. Χρειάζεται ε, ένας ακόμα ίδιος πόρος για να χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί από το Ρούσβελτ στο Τραμπ είχαμε ε, φόρο 38% επί των κερδών και στην Ευρώπη πέσαμε στο 19%. Και στον, με τον Τραμπ, παρόλο που έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις, ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων είναι στο 24%. Πάνω από το 19% που έχουμε εμείς. Χρειαζόμαστε ίδιους πόρους, χρειάζεται η, η το Κοινοβούλιο να ε, συμφωνήσει στα θέματα αυτά, όχι μόνο η Επιτροπή Προλογισμών, όχι μόνο η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Πρέπει να σας πω πως χρειαζόμαστε ένα πραγματικό σχέδιο ε, για την συνανάπτυξη με τις χώρες του Νότου μέσω της έρευνας. Ξέρουμε πως υπάρχουν λύσεις, αλλά αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Green Deal, δεν θα πρέπει να περικόπτουμε τον προλογισμό, πρέπει να επενδύουμε όλο και παρατηρήσουμε πάνω για κάθε χωριό, για κάθε οικογένεια, για κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση θα πρέπει να τους πούμε πως όταν κάνουν κάτι υπέρ του περιβάλλοντος το κόστος θα το αναλάβουμε εμείς συλλογικά έτσι ώστε να καταφέρουμε να ε, είμαστε στο μηδενικό, στις μηδενικές εκπομπές ή ακόμα καλύτερα τώρα για το φόρο στην κεροσύνη να σας πω τι έκανε ο Μπαράκο Ομπάμα. Είχε ε, τον νόμο ΦΑΤΚΑ που είπε καμία τράπεζα δεν θα ε, εργάζεται στις Ηνωμένε Πολιτείε αν δεν έχει απόλυτη διαφάνεια προς την Αμερικανική εφορία. Έγιναν πάρα πολλά ε, για τα θέματα της κατηγοροποίησης και την ταξονομία και μπορούμε να πάμε λίγο παραπάνω έτσι ώστε καμία ασφαλιστική εταιρεία, καμία τράπεζα να μην μπορεί να εργαστεί στην Ευρώπη αν δεν είναι απόλυτα διάφανη οι λογαριασμοί της και με τον τρόπο αυτό να χρηματοδοτήσουμε τον Green Deal σύμφωνα με το όσα είπαμε στο Παρίσι για να κερδίσουμε τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος. Και να σας πω πως αυτή τη βδομάδα ε, γιορτάζουμε ε, την γέννηση του άνθρακα και του χάλιβα της κοινότητας αυτής ε, που ήταν η απαρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας θυμόμαστε τα λόγια του Ρόμπερτ Σούμαν που είπε πως η παγκόσμια ειρήνη ε, θα διατηρηθεί μόνο αν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ειρήνη. Και αυτά τα είπε ο Ρόμπερτ Σούμαν και θα τα γιορτάσουμε σε δύο εβδομάδες. Γιατί αν δεν καταφέρουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μεθαύριο να αλλάξουν το παιχνίδι, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μοιάζει να θέλει να το κάνει, τότε εμεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μα, να φέρουμε καινούριε ιδέε στο τραπέζι και να αλλάξουμε το παιχνίδι ριζίκα. Είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Το πάθο ξεπερνάει προφανώ τον προπολογισμό του 2021 ω θέμα. και μπορούμε να εντάξουμε αυτό το σημείο στις γενικότερες ανησυχίες που θέλουμε να συζητήσουμε. Όταν λέτε ότι πρέπει να μειώσουμε ε, τουλάχιστον στο μισό τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, εννοούμε ότι δεν θέλουμε να τις μειώσουμε στο μισό σε σχέση με το 1990, Σημαντικό να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν είναι ακριβώς η ίδια προσπάθεια. Λοιπόν, ερωτήσεις. Δεν έχω κάποιον από το ΕΛΚ. Ξεκινάμε με τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες, κυρία Γκούτλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή για την ε, παρουσίαση αυτή και την προθυμία του να έχουμε μια εύρυθμη συνεργασία μεταξύ της δικής σας Επιτροπής και της δικής μας. Έχουμε ήδη κάνει μια καλή αρχή για να έχουμε έναν καλό διάλογο μεταξύ μας. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Μπένοβα Τη δικιάς μας ε, και οδού εισηγήτρια που δεν μπορούσε να είναι εδώ και θα πω κάποια λόγια εκ μέρου της. Προηγουμένως, ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλη την παρουσίαση. Πραγματικά την ε, εκτίμησα θα θέλατε το Κοινοβούλιο να αναλάβει υπεύθυνη δράση κάνοντας ένα μεγάλο βήμα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για ολόκληρο τον κόσμο για όσα συμβαίνουν γύρω μας και προκειμένου να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για μια σταθερή και βιώσιμη για το μέλλον οικονομία έχοντας κατά νου και την ε, Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal. Πραγματικά ήταν εμψυχωτικό να σας ακούει κανείς. Και μιλώντας εκ μέρους της κυρίας Μπένοβα, να πω ότι και εκείνη είναι αναφανδόν υπέρ της έκθεσής σας. Υπάρχει σοβαρή στήριξη. Χαιρόμαστε που οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων βρισκόνται πραγματικά στο επίκεντρο της δουλειάς σας και θεωρούμε ότι στον προπολογισμό το 2021 πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, οδεύουμε προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και για την βιοπικιλότητα και τον στόχο δαπάνης του 10% αυτό για μας είναι σοβαρής. Είναι μεγάλη σημασία. Επίσης η καταπολέμηση του καρκίνου είναι κάτι που θέλουμε να το δούμε να ενισχύεται στον προπολογισμό εκ μέρους της ομάδας μου, να τονίσω και τη σημασία του να έχουμε και επαρκείς πόρους για την Πράσινη Συμφωνία. Δεν χρειάζεται εδώ να επιμείνω, ακούω πώς επιμένετε εσείς από μόνος σας. Ενθαρρυντικό αυτό. Δεν θέλουμε να είναι απλώς ένα συγχώρο χάρτη για την Ευρώπη η Πράσινη Συμφωνία. Θέλουμε να λειτουργήσει πραγματικά να είναι δραστική και θέλουμε να έχουμε απαραίτητους πόρους για να γίνει η μετάβαση. Αυτή είναι για μας η προτεραιότητα. Πιστεύουμε ότι το, ο προπολογισμός το 2021 είναι το πρώτο λιθαράκι για την ε, πολιετή δημοσιονομική περίοδο μέχρι το 2027. Έχουμε προεδρικές εκλογές τα ερχόμενα χρόνια και θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά ε, επιτυγχάνουμε να γίνει μια μετακίνηση, μια πραγματική καμπή για την Ευρώπη. Και φαντάζομαι ότι περιτεύει να σας το διευκρινίσω, αλλά η δίκαιη μετάβαση ε, είναι σημαντικό. Πρέπει να καταστεί εφικτή. Το είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας. Και επίσης, απλώς να πω ότι θα υποβάλουμε τροπολογίες για το σημαντικό ε, υγειονομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Θα δείτε τα σχετικά από εμά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προθυμία σας, το πνεύμα συνεργασίας που επιδεικνύεται και για την παρουσίαση που μόλι κάνατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για το ΕΛΚ, η κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ. Δεν εκπροσωπώ το ΕΛΚ, αλλά τον εαυτό μου διότι ο κύριος Λίζα δεν βρίσκεται εδώ. Δεν ζήτησε το λόγο, οπότε είστε η μόνη εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περίοδου. 2000, το 2021 είναι συμβολικό έτος ως προς αυτή την έννοια. Θέλω να Παναλάβω την τοποθέτηση τη ομάδα μου σε σχέση με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Για μα είναι σημαντικό να έχουμε κάποιο περιθώριο, χρονικό περιθώριο ε, για να βρούμε το σωστό προπολογισμό παρά να έχουμε ντε και καλά συμφωνία αύριο μεθαύριο και να μην είναι αρκετά φιλόδοξο ο προπολογισμό επειδή βιαστήκαμε. Ε, Ω προ του πόρου και την εφαρμογή τη Πράσινη Συμφωνία, θέλω να ρωτήσω για την εφαρμογή του μηχανισμού δίκαιη μετάβαση. Πώ το έχετε φανταστεί, πώ θα σχεδιαστεί και ε, υπολογίζετε να λειτουργήσει πραγματικά ο μηχανισμό αυτό και να φέρει αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Δεν έχω κάποιον ε, ομιλητή από την ομάδα ID για τους πρασίνους. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Απλώς ένα σχόλιο για αυτά που υπόθηκαν. Δηλαδή περισσότερο να εκφράσω μια ανησυχία δική μου. Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε να λέμε για φόρο ε, για το κρέας, φόρο για, τα, ε, για τη ζάχαρη, φόρο για τα καύσιμα, φόρο για ένα σωρό πράγματα. Συμφωνώ ότι τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται και πρέπει η φορολόγηση να είναι ισότιμη μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει ούτω ή άλλω, όχι σε σχέση με το τι κάνουν οι ΗΠΑ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά. Είναι κάτι που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Η ανησυχία μου όμω είναι ότι όλοι αυτοί οι φόροι για να πάρουμε πόρου ε, που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσει η Πράσινη Συμφωνία είναι κάτι που θα επιβαρύνει τελικά του πολίτε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, λοιπόν. Και μιλήσατε και για την Συμφωνία ΕΚΑΧ ε, των ε, θεμελιωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πρωτοειδρύθηκε. Ναι, η ενέργεια είναι κάτι σημαντικό για να προχωρήσουμε και σήμερα όπω ήταν και τότε. Όμω τότε οι ιδρυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φρόντισαν να γίνει Ενεργειακή Ένωση τιμωρώντα και επιβαρύνοντα του πολίτε. Ε, οι τιμέ ε, του Χάλιβα και του Άνθρακα ε, πέρασαν υπό έλεγχο, αλλά όχι βάζοντα το υπερβολικό κόστο να το πληρώνουν οι πολίτε. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάμε τι είναι αυτό που μπορεί να λειτουργήσει τιμωρητικά για τι πιο ευπαθεί ομάδε, τι πιο αδύναμε ομάδε του πληθυσμού μα. Και αυτό να μα απασχολήσει πρωτίστω. Ευχαριστούμε. Για τους πρασίνους ο κύριος Έκχαουτ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο α, για την παρουσίασή του, τη διεξοδικότατη παρουσίαση και επίσης που καταδείξατε τη συμφωνία του να δείξουμε πόσο σημαντικός είναι ο προπολογισμός για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Διότι αυτή είναι η συζήτηση που τίθεται για το 2021. Τελικά έχουμε περάσει ήδη στη συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που τώρα μα απασχολεί. Πραγματικά λοιπόν, ό,τι πούμε ω Ευρωκοινοβούλιο για τον προπολογισμό το 2021 θα σημαδέψει και το τι ε, θα αποφασίσει το Συμβούλιο για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ δεν είμαι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή την εβδομάδα. Και αν δω τι προτάσει του κυρίου Μισελ, πραγματικά ελπίζω όντω να μην ολοκληρώσουν αυτή την εβδομάδα γιατί εκεί βλέπει κανείς ακριβώς τι συμβαίνει. Όλα τα καινούρια, ε, οι νέες και ρεξικέλευτες ιδέες ε, μικραίνουν όλο ένα και περισσότερο στη χρηματοδότηση που λαμβάνουν. Γιατί χώρες όπως η δική μου δεν θέλουν να πληρώνουν πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της συνοχής ε, κοιτάζουν να προσπιστούν τα δικά τους συμφέροντα, την γεωργική πολιτική και μετά η καινοτομία, η πράσινη συμφωνία και αυτά όλα ένα συρρυκνώνονται. Εκεί λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε, να πατήσουμε πόδι και να το εμποδίσουμε και εκεί έρχεται και κολλάει η παρουσία Πραγματικά λοιπόν πρέπει να περάσουν ισχυρά μηνύματα και θέλω να ευχαριστήσω ε, τον πρόεδρο για το σχέδιο, γιατί πραγματικά ε, θα μπορούσε να ενδυναμωθεί. Δεν έχουμε ποσοστό που να αναφέρεται συγκεκριμένα για το τι θα αποδώσουμε στο κλίμα, λόγου χάρη. Και οι αριθμοί που αναφέρατε εσεί δείχνουν πόσο σημαντικό είναι ήδη αυτό το θέμα. Ο κ. Μισελ και εκεί πραγματικά είναι πολύ επιφυλακτικό, ε, πολύ αδύναμα αυτά που προτείνει. 25% αλλά δεν είναι και πολύ δεσμευτικό. Είναι μία σύσταση, μία συμβουλή για το τι θα έπρεπε να γίνει. Εάν λοιπόν αφήσουμε το Συμβούλιο να απομακρυνθεί από αυστηρούς δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα, ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το εμποδίσουμε, διότι η Επιτροπή μας είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ούτως ή άλλως προηγουμένως για τη βιοπικιλότητα. Ε, ο κύριος Μισελ το ανέφερε μεν και δείξατε πόσα όλα, πόσο όλα είναι αλληλένδετα σε σχέση με την επικοινότητα. Εμείς θελήσαμε να υπάρξει εδώ πρόσθετη χρηματοδότηση σε σχέση με τους στόχους ε, αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Αυτό έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο στην σχετική του, στο σχετικό του ψήφισμα. Όμως αυτό που αρχίζει και γίνεται πολύ σημαντικό είναι το πώς θα ελέγχουμε την επίτευξη των κλιματικών στόχων, το climate proofing όπως λέγεται. Δηλαδή, ε, πρώτον να αποδώσουμε όσα θέλουμε στους κλιματικούς στόχους, αλλά μετά να κοιτάζουμε ότι δεν είναι και επιζήμια αυτά που έχουμε προβλέψει ως προς το κλίμα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τέτοια νομοθεσία που να βεβαιωθούμε ότι ε, αποφεύγουμε και τον αρνητικό αντίκτυπο κατά τις πράσινες συμφωνίες και του επίτευξης των κλιματικών μας στόχων. Ε, εκεί χρειαζόμαστε την κατάλληλα εργαλεία. Και οι τροπολογίες μας σκοπό έχουν να ζητήσουν όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζητά υποβολή εκθέσεων και λογοδοσία σε σχέση με το πρασίνισμα, το κάνει με τον πιο επιφανειακό τρόπο. Δηλαδή, ξέρουμε τι κάνει στη Γεωργία για το κατά πόσον ε, οι επιδοτήσει χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Ε, το ποσοστό του πρασινίσματο δεν υπολογίζεται σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάμε όταν μιλάμε για τα ποσοστά αυτά, να κοιτάμε τι είναι πραγματικά πραγματικά πρόταση πρασινίσματο, τι πάει στο κλίμα τη, στη βιοπικιλότητα και να υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί. Θα το συμπεριλάβουμε αυτό στην τροπολογία μα και θα φροντίσουμε να σα ε, οθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση με τις προτάσεις μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην Επιτροπή μας να φανεί ότι θέλουμε να πάρει σάρκα και οστά το όλο εγχείρημα της Πράσινης Συμφωνίας και να γίνει ε, μια πραγματικότητα που θα ωφελήσει πραγματικά την Ευρώπη συντηρήθηκε με μεταρρυθμιστέ. Panie Przewodniczący, Panie e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ε, ξεκινήσατε τη συζήτηση αυτή με την παρουσίασή σας. Βλέπουμε πώς ε, συγκινήσεις και έντονα αισθήματα προκαλεί αυτή η προοπτική του πολιτικού προπολογισμού. Ελπίζουμε πραγματικά να γίνει και πράξη. Ξέρουμε ότι έχουμε πει μέχρι το 2030 πρέπει να φτάσουμε σε 40% μείωση των ε, εκπομπών. Αυτό δεν θα το πετύχουμε, το ξέρουμε και ίσω να πετύχουμε το 36%. Και με το Brexit μιλάμε πλέον για 34% και αν. Ε, έτσι λοιπόν ε, όταν κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις φιλοδοξίες του σε συγκεκριμένα προγράμματα και απτά μέτρα ε, και συγκεκριμένους στόχους, αυτό συμβαίνει. Εκεί λοιπόν ανησυχούμε σε σχέση με το Συμβούλιο, διότι είναι γεγονός ότι εδώ για την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι σαφές. Ε, εμείς τα γνωρίζουμε τα του κλίματος και του, της βιοπικιλότητας και ξέρουμε πως αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε οικονομικούς όρους. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται σε κράτη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η... Ε, αλλού. Και όταν ακούει κανείς ε, μιλά για φόρους, πρέπει να κοιτάξει πού ε, θα πληρωθούν όλα αυτά. Θα πρέπει τους πολίτες να μπορούμε να τους πείσουμε, να τους ε, εξηγήσουμε ότι ότι πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για το νερό, για το ηλεκτρικό, για την διαχείριση των λιμάτων και ούτω καθεξής. Πρέπει κάπως να το πείσουμε. Ε, άκουσα λοιπόν την παρουσίαση του συγητή, ήταν ε, πραγματικά γεμάτη ενθουσιασμό. Όμω θα πρέπει και να κοιτάξετε να κάνετε και συγκεκριμένου υπολογισμού, με συγκεκριμένου αριθμού και ποσοστά. Θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποια στιγμή τα κράτη-μέλη να έχουν υπολογίσει στο χαρτί με συγκεκριμένα ε, ψηφία του αριθμού που θέλουν να πετύχουν διότι εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για 55%. Θέλουμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ποσά και συγκεκριμένες αποφάσεις. Όταν είναι κανείς υπουργό οικονομικών κάποιου κατούς μέλους ε, και έχει μια συγκεκριμένη απόφαση που μπορεί να μην αρέσει, πρέπει να βρει και μια πηγή χρηματοδότηση, τουλάχιστον για μια δεκαετία. Εδώ εμείς μιλάμε για μια επταετία. Ε, οπότε, ε, αυτό που καταρχάς θέλω να σας ζητήσω είναι να κοιτάξετε να αναλύσετε πολύ προσεκτικά τι μπορεί να γίνει, τι είναι απαραίτητο σε κάθε κάτω μέλος, ώστε να μιλήσουμε πια για συγκεκριμένες απτές λύσεις. Ο κύριος πρόεδρο, ο, πρόεδρος μας βρέθηκε στην συνεδρίαση όπου ο κύριος Τίμερμανς και ο Επίτροπος για τον Προπολογισμό ε, μιλήσανε πολύ θεωρητικά για όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουν από πού θα προέλθουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε για τον ε, επτάετη προπολογισμό μας. Πού θα βρεθούν τα 7 δις, τα 5 συν 2 δις, θα είναι ε, από κάπου αλλού, από τον προπολογισμό, ε, θα είναι τελείως καινούρια. Και επίσης, τι θα κάνουμε για να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσεις, τις επενδύσεις των ιδιωτών. Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα, ένα τέτοιο περιβάλλον, ώστε η Πράσινη Συμφωνία πραγματικά να φαίνεται και ρεαλιστική και βιώσιμη. Ευχαριστούμε για την Ιγκού, ο κύριος Κόκαλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετική η δουλειά που κάνατε. Η πιο πιεστική πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι ο πλανήτης μας και ο κόσμος μας να μείνουν υγιείς. Αυτό είναι το βασικό και η απάντηση που δώσαμε είναι το Green Deal. Τώρα, αυτά ζητάει η Κομισιόν και ψάχνει ο εισηγητή συμμαχίε από την Επιτροπή μας που είναι η Επιτροπή για το Περιβάλλον. Εμείς προτείνουμε στον προπολογισμό του 2021 να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να εφαρμόσουμε το Green Deal. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε σταδιακά βήματα. Θα πρέπει να δυναμητήσουμε την κατάσταση με δημοκρατικό τρόπο και ακολουθώντα το χρονοδιάγραμμα τη επιστήμης. Γι' αυτό είπαμε 100 ημέρε. Ίσως τα δέκα χρόνια φτάνουν για να βάλουμε κάποιον στην, ε, στον πλανήτη Αφροδίτη. Πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός να είναι ο πρώτος που θα βάλει ε, το περιβάλλον στην κορυφή και θα κάνει ένα κβαντικό άλμα προς την κατεύθυνση της επιδίωξης των στόχων μας. Στηρίζουμε τον εισηγητή και στηρίζουμε το 1,29 ε, του ΑΕΠ στον επόμενο προπολογισμό και για την πρόταση του Προέδρου της, ε, ε, του Συμβουλίου ε, για τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να το απορρίψουμε και να στηρίξουμε τον εκπρόσωπό μας βασιζόμενοι στο σχετικό άρθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω και μία ερώτηση για σας για το 1,63 από τα ΕΚΤ και τα 240 δις ε, για την αγορά ομολόγων. Γιατί να μην κάνουμε, για να μην παρουσιάσουμε λοιπόν, κάποια ομόλογα πράσινα ε, στα πλαίσια του Green Deal. Τρεις ομιλητές έχω ακόμα και εγώ είμαι στον κατάλογο και μετά θα έχετε και 10 λεπτά για να κλείσετε το θέμα. Πίτερ από το Άλκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Συγγνώμη που έχασα την παρουσίασή σας, την παρουσίασή σας αλλά είχαν λυμμένες υποχρεώσεις. Το είπε και ο κύριος Έκχαουτ. Η συζήτηση σήμερα έχει άμεση σχέση με τα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και θέλω να πω και εγώ δύο-τρία πράγματα σχετικά. Ο κύριος Μισελ έριξε κάποιο φως σε κάποιες υποθέσεις, αλλά και αρκετές σκιές. Ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου φαίνεται να δέχεται το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης και υπάρχει κάποιο σχετικό άνοιγμα για ιδίους πόρους. Επίσης για να φόρο των πλαστικών για το σύστημα ανταλλαγών, ε, δικαιωμάτων ανταλλαγών αερίου του θερμοκηπίου, το ETS. Θα δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Και θα δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε και στο μεταγενέστερο διάστημα, αν θα μπορούμε να δεχτούμε την έκβαση του Συμβουλίου ή όχι. Γιατί σχετική περικοπή στην έρευνα είναι απαράδεκτη αυτή για την προοπτική για την ε, Επιτροπή μας. Θέλουμε να, να συνεχιστεί ο αγώνας κατά του καρκίνου. Θέλουμε να υπάρξει καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Αυτά έχουν όλα άμεση σχέση με την έρευνα. Το 33% που προτείνεται από τον κύριο Μισελ δεν φτάνει. Και σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας είναι εντελώς απαράδεκτο το Εράσμους να έχει τέτοια κακή χρηματοδότηση. Και μια παρατήρηση για, τον συνάδελφο από τις, για τη συνάδελφο από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Το 40% δεν είναι ορθό. Το 40% θα το πετύχουμε έτσι καλλιώ και αν τα κράτη-μέλη δεν έχουν μπει στο σωστό δρόμο, θα πρέπει να τα ε, επαναφέρουμε στην τάξη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και από το 40% και ίσως και περισσότερο από το 50% να πετύχουμε βάσει των αναλύσεων τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα δούμε. Πάντως, αυτό που φρονώ είναι ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό εδώ. Συζητούμε για ποσά μεταξύ του 1 και του 1,3% του ΑΕΠ. Δηλαδή ε, όλος, όλη η συζήτηση γίνεται για το 1,0 ή το 1,1 στο Συμβούλιο ή το 1,15. Δεν είναι τίποτα παραπάνω, κανένα μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή το 98 και παραπάνω του κρίματος που κυκλοφορεί στην Ευρώπη δεν έχει καμιά σχέση με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εκεί είναι που μας λείπει η χρηματοδότηση και γι' αυτό θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα στου εθνικούς προπολογισμού και κίνητρα στην ιδιωτική οικονομία, την οικονομία των ιδιωτών για να ενισχύσουμε τη θέση μας, για να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για το δεξίδιο του άνθρακα και τι τιμές μπορούμε να επιβάλλουμε εκεί που δεν υπάρχουν ε, για το παράγουν τέτοιους ρήπους, να δουν πώς μπορούν να τους περιορίσουν και επίσης να ελαφρύνουμε λίγο τη θέση όσων προτείνουν νέε τεχνολογίες λύσεις απαλλαγμένες από το διοξείδιο του άνθρακα και θα μπορούσαν οι τιμές τους να ε, ενισχυθούν, ε, να μην είναι τόσο υψηλές δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώ θα ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό υπολογισμό, εάν καταφέρουμε να προσελκύσουμε και τι σχετικέ ιδιωτικέ επενδύσει. Ευχαριστούμε σοσιαλιστές και δημοκράτες ο κύριος Λουένα. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αγαπητέ συνάδελφε για αυτή την καταπληκτική παρουσίαση που κάνατε και για το ότι υπερασπιστήκατε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για συμβιβασμού. και Κάναμε συζητήσεις, κάναμε διαπραγματεύσεις. Τώρα έφτασε η στιγμή ε, να συζητήσουμε τα καυτά θέματα και θα ξεκινήσω εγώ με το φορολογικό. Ξέρετε τα κίτρινα γυλαίκα και τι κάνουν. Κανείς δεν θα ήθελε αν δεν εξηγήσουμε τις αναγές που πρέπει να γίνουν να έχουμε προβλήματα κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έχουμε εντάξει τον παράγοντα δίκαιη κατανομή ευθυνών και βαρών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Γιατί όταν στην ιστορία της Ευρώπης ξεκίνησε το κράτος πρόνοιας, ξεκίνησε γιατί είπαμε θα πρέπει το κέρδος να συνεισφέρει περισσότερο στην στήριξη των Άρα λοιπόν δεν θα μπορεί να αποτελεί ένα απλό χανζαπλάστ ε, ή ε, περιβαντολογική φορολογία. Θα πρέπει με γεωγραφικό τρόπο, γιατί μιλάμε για το Νότο και το Βορρά, το είπε και ο συνάδελφος του ΕΛΚ που μίλησε για τις συνεισφορές, να βρούμε έναν τρόπο να είναι η κατανομή δίκαιη. Και η συζήτηση, ε, όταν έχουμε τέτοιες τεράστιες ε, αλλαγές στην κοινωνία, πάντα περνά από το θέμα του φορολογικού. Επίσης, θα μιλήσουμε λοιπόν για τις ΑΠΕ οι οποίες βοηθούν στη μείωση των εκπομπών σε ποσοστό πάνω από 30% και θα πρέπει να παίξουν ρόλο. Αυτό που ζητώ εγώ εδώ είναι να αυξήσουμε ε, επίσης και να αυξηθούν τα κονδύλια στο ε, προπολογισμό για το σχέδιο δράσης για τη μάχη κατά του καρκίνου. Αυτό είναι ένα ακόμα δικό μου αίτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Λαρού για την παρουσίασή του και πρέπει να πω ότι και από δική μου πλευρά Πραγματικά, αν ψάχνατε συμμάχου, να, εγώ είμαι δικιά σα. Πραγματικά η εκκλησία σα με ευαισθητοποιεί και συμφωνώ με πολλά από αυτά που προτείνετε. Διότι φρονώ ότι σε αυτή την ιστορική στιγμή όλοι πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε δημιουργικά, ε, εφάνταστα και λίγο out of the box. Να κοιτάξουμε δηλαδή, να βρούμε λύσει εναλλακτικέ. Έχουμε μπροστά μα τεράστιε προκλήσει και δυσκολίε. Πρέπει λοιπόν και περισσότερο να εργαστούμε και σκληρότερα και με ε, πνεύμα δημιουργικό. Ε, γι' αυτό λοιπόν πραγματικά Ωραία τα είπατε με το fact ε, κλίμα ε, και το τι κάνουν οι τράπεζες λόγω χάρη στην Ευρώπη, εάν υπάρχουν επενδύσεις, ορυκτά καύσιμα ή όχι, όλα αυτά είναι σημαντικά και η έκκλησή σας για να βεβαιωθούμε ώστε όλα τα κονδύλια που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλέ φορέ καταλήγουν στην κερδοσκοπία, θα πρέπει να πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία και σε δράσει προστασία του περιβάλλοντο και τη βιοπικιλότητα. Εκεί θα προσυπογράψω πλήρω και πρέπει να, να αναλάβουμε τολμηρή δράση, διότι μιλάμε για την Πράσινη Συμφωνία. Μα χρειάζεται ακριβώς μια πραγματική. Ε, ε, ε, πράσινη συμφωνία, ώστε να είμαστε αξιόπιστοι ω Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ, τα είπατε κι εσεί. Τα είπατε κι εσεί οι υπόλοιποι συνάδελφοι σε σχέση με τι προτάσει που έχουμε επιτάπητο στο Συμβούλιο. Και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πάψουμε να είμαστε σε επιφυλακή. Θα είναι πραγματικά μία ε, ανταλλαγή αρκετά έντονη γιατί θέλουμε ο προπολογισμό του 2021 να είναι στο ύψο των προσδοκιών μα. Κάποιε μικρέ παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα για του ιδίου πόρου. Το έθεξαν πολύ. Εγώ ε, πραγματικά θέλω να επαναλάβω μια ιδέα, μια πρόταση, εδώ, καινοτόμα, ρηξικέλευθε ίσως, ε, που θα μπορούσε να επιτρέψει ε, ένα εισόδημα για το Ευρωπα... Ευρωπαϊκής... προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Λέγεται φόρο για τις πρόσθετες εκπομπές. Η ΜΕΑ έχει ονομαστεί. Θα επιβληθεί στα σύνορα και θέλει να προστατεύσει τις εταιρείες που εργάζονται αποκλειστικά στην Ευρώπη. Δηλαδή για, την, για τον ΦΠΑ για το ΦΠΑ θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση σε σχέση με το περιεχόμενο σε άνθρακα που έχουν τα προϊόντα και ότι προκύπτει από τι επιχειρήσει μα. Εκεί θα πρέπει να προστατεύσουμε επιχειρήσει και εταιρείε που έχουν παραγωγή πολύ καθαρότερη, απαλλαγμένη από άνθρακα σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόσθετο φορό από αυτού που ψάχνει η Ευρώπη. Επίσης δεν αναφέραμε και εδώ είναι κάτι που θα ε, πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε θεωρώ Πολλά κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κάνουν τι απαραίτητε επενδύσει για το περιβάλλον και το κλίμα και πρέπει να αναθεωρήσουμε του κανόνε οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει επιτέλου να δούμε το κατά πόσον έχουν κατανεμηθεί σωστά τα κονδύλια στα πλαίσια του Συμφώνου ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης προς τον κοινωνικό κυρίως πυλώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ως εισηγητής για την έκθεση Envy θα ολοκληρώσω την όλη ανταλλαγή πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή μας στα γαλλικά. Δεν θα φορολογήσουμε τους πολίτες. Μιλώ πολύ ε, γρήγορα, αλλά δεν είναι αυτό που επιθυμώ. Κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία, 30%. Ε, και υπάρχουν Γάλλοι και Πολωνοί και Γερμανοί που δεν έχουν ένα ευρώ στην τσέπη κάθε μήνα. Δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε. Είναι οι ευάλωτοι. Δεν θα πληρώσουν αυτό το λογαριασμό δίκαιη μετάβαση, ε, τότε και δίκαιη φορολόγηση και μαζική χρηματοδότηση και όχι μόνο για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τον άνθρακα, δίκαιη χρηματοδότηση και με αυτό θα συνταχθεί όλη η Ευρώπη και νομίζω ότι και οι Ισπανοί ε, υπουργό ε, και ο Βέλγος όταν έρχονται οι Πολωνοί υπουργοί στην ε, Ευρώπη μας λένε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Λοιπόν, δίκαιη μετάβαση, δίκαιη και μαζική χρηματοδότηση για να επανακινήσουμε την Ευρώπη τον 27 και αν όχι τον 27 τον όσον το δυνατόν περισσότερο κρατών μελών. Δώστε μου δύο λεπτά ακόμα και τελειώνω. Τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών για το χρονοδιάγραμμα σας τα είπα το 1,7 που μας ε, πρότειναν, ε, κόψαν την έρευνα, δεν έχει τίποτα για το κλίμα. Ε, δεν το λες και σοβαρή πρόταση. Όχι, θα πούμε. Και θέλουμε λίγο χρώμα ακόμα για να παρουσιάσουμε τις δικές μας προτάσεις ως Κοινοβούλιο. Για τις νέους σπόρους τα είπα. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Στόχος μου ήταν να σας πω δεν θα δουλέψει μόνη της η Επιτροπή Προπολογισμών. Θέλουμε και εσάς να μας βοηθήσετε. Θέλουμε την πραγματογνώμη, το γνωμοσύνη σας και την νομική βάση να τη βρούμε. Γιατί αν ε, καταφέρουμε να απεμπλοκάρουμε τη χρηματοδότηση και μετά μας πούνε ξέρετε πολύ ωραία όλα αυτά, συμφωνήσετε το νούμερο, αλλά νομική βάση δεν έχετε, θα το πετάξουμε στον κάτω των αχρήστων. Οπότε παρακαλώ πολύ ε, να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίες, πού μπορούμε να στείλουμε αυτά τα κονδύλια, τι είναι το καινούριο που μπορούμε να φέρουμε. Ευρωπαϊκή ειναι το καινουργιο που μπορουμε κάντε τη δουλειά σας. Βρείτε νέους πόρους, μέσω προϋπολογισμού, εκτός προϋπολογισμού, Ο καθένας ό,τι μπορεί για να βοηθήσει ποια σχέδια χρειαζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε, ποια είναι η νέα νομική βάση και να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτή τη στιγμή τον προϋπολογισμό τη στιγμή της εκταμίευσης. Τρία-τέσσερα χρόνια θα χρειαστεί. Γιατί κάποιο θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Κάποιο θα έχει καλή χρηματοδότηση, κάποιο θα έχει καλύτερη νομική ε, βάση. Ευχαριστώ όλους και όλες. Λείπει ο Πρόεδρος, ας συνεχίσουμε παρόλα αυτά. Και να δούμε το επόμενο σημείο. Έχουμε τον έλεγχο καταλληλότητας για την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τόσο παθιασμένη η συζήτηση προηγουμένη ε, για το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Green Deal θα έχει τους κατάλληλους πόρους. Χαίρομαι που μπορούμε να επιστρέψουμε σε ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή αν είμαστε σοβαροί και αν απλώς δεν ε, ε, ε τηρούμε τα προσχήματα για το περιβάλλον. Έλεγχος καταλληλότητας το Νοέμβριο που βασίστηκε σε μια ενδελεχή εξέταση των δεδομένων που έστειλαν για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα από το 8 μέχρι το 18 που έστειλαν όλα τα κράτη-μέλη. Δεκαετία ολόκληρη η οποία μελετήθηκε λεπτομερώς και έχουμε και όλο το feedback από τους ενδιαφερόμενους. Κάναμε και μία σειρά από μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων 7 κράτη-μέλη και ο τρόπος που αυτά ε, εφαρμόζουν την νομοθεσία. Βουλγαρία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Σλοβακία ήταν οι 7 τυχεροί. Και κάναμε και μια εξαιρετικά ενδελεχή εξέταση της βιβλιογραφίας, πάνω από 600 πηγές τεκμηρίων, με ε, μοντέλα υπολογιστικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να ε, ε, διεξάγουμε τα συμπεράσματα από αυτές τις αναλύσεις. Καταλήγουμε λοιπόν πως η πολιτική αυτή σε γενικές γραμμές είναι επιτυχημένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε λύσει το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Ευρώπη. Το αντίθετο μάλιστα. Γνωρίζουμε όλοι πως μέχρι και σήμερα 400.000 περίπου πρόοροι θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στην κακή ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Την τελευταία δεκαετία έλαβαν χώρα αρκετές προσπάθειες, μπορώ να το πω αυτό, και ο αριθμός των πρόωρων θανάτων που είχαμε πριν από μερικά χρόνια ήταν περισσότεροι γιατί έφταναν το 1 εκατομμύριο περίπου πολίτες. Άρα λοιπόν κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα είναι υπερβολικά υψηλός ο αριθμός των προώρων θανάτων. Συμπεράσματα. Τέσσερις βασικές κατηγορίες συμπερασμάτων. Μπροστά μας να τα δούμε. Με το δίκτυο που δημιουργήσαμε των 4.000 σταθμών μετρήσεων που ακολουθούν κοινά κριτήρια, έχουμε κάνει κάτι το πετυχημένο. Αναγνωρίζοντας βέβαια στον έλεγχο καταλληλώτες πως αυτά τα δίκτυα παρακολούθησης μπορούν να βελτιωθούν παραπάνω για να έχουμε ακόμα πιο αξιόπιστα και συγκρίσιμα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις και των 27 κρατών μελών. Uh, Η νομοθεσία Επίσης, έχει εισάγει ξεκάθαρα πρότυπα για 13 εξαιρετικά επιβλαβείς ρηπογόνες ουσίες για τον άνθρωπο. Και τα επιστημονικά τεκμήρια έχουν επιβεβαιωθεί και αναγνωρίζουμε πως το επίπεδο των προτύπων σήμερα δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει δώσει ο ΠΟΗ για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. Αναγνωρίζουμε πως γενικά οι οδηγίες οι οποίες διευκόλυναν την διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των αντικειμενικών και συγκρίσιμων δεδομένων έτσι ώστε να μεταβούμε στην πλήρως ψηφιοποιημένη εποχή σημαίνουν πως θα χρειάζεται τον τρόπο αναφοράς να τον βελτιώσουμε ακόμα παραπάνω με καλύτερα μοντέλα και προβλέψεις, με καλύτερη παρουσίαση των δεδομένων, με καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και των όσων χαράσουν πολιτική επιτόπου. Και τέλος, τελευταία κατηγορία συμπερασμάτων έχει να κάνει με το γενικά οι οδηγίες αυτές μόνο μερικούς, έχουν ε, σεβαστεί το στόχο μας που είναι να αντιστρέψουμε τα αποτελέσματα, τα αρνητικά, τις αρνητικές συνέπειες της κακής ε, ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα, γιατί 20 κράτη-μέλη ακόμα αναφέρουν ε, τιμές παραπάνω από τα δικά μας όρια τα ευρωπαϊκά και αυτό έχει να κάνει με το πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες σε εθνικό επίπεδο και να συμμορφωθούν με την ένταξη αυτών των προτύπων ε, στην νομοθεσία περί περιβάλλοντος μεταφορών και γεωργίας σε εθνικό επίπεδο. Καταλήξαμε λοιπόν στο fitness check πως σε γενικές γραμμές είναι κατάλληλη νομοθεσία αυτή. Παράλληλα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε λοιπόν τα 7 κομβικά διδάγματα Πρέλουμε πιο αυστηρές πρόνοιες για την παρακολούθηση και να αναθεωρήσουμε τα πρότυπα έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στις τάσεις του ΠΟΗ. Και πρέπει να σας πω πως εκεί συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους και αναθεωρούμε τις συστάσεις 2006 έτσι ώστε νέες συστάσεις να εκδοθούν ελπίζουμε το 2021 και ξέρετε κι εσείς πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει πως το 2021 θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης μηδενικής ρήπανσης για τον ατμοσφαιρικό αέρα, για τα εδάφη και για τα ύδατα. Με χαρά θα ακούσω και τις δικές σας απόψεις για αυτό τον έλεγχο καταλληλότητας και βασιζόμαστε στη δική σας δημιουργικότητα. Κάποιος είπε προηγουμένω πως είναι σημαντικό να είναι κανείς δημιουργικός, να σκέφτεται κανείς εκτός των τετριμένων, out of the box και να καταφέρουμε αυτό το μηδέν ε, της εκατορύπανσης με βιοπικιλότητα και με ένα υγιές περιβάλλον για την Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Για το ΕΛΚ, η κυρία Σνάιντερ, ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με όσα είπατε. Μιλήσατε για το 2004 και τη διαδικασία παρακολούθησης από τότε, αλλά εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε λίγο την ατμόσφαιρα και για την αποδοχή της οδηγίας και γενικότερα για τα πρότυπα που ισχύουν. Το θέμα είναι λοιπόν τι συγκεκριμένε και προτάσει έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση υλοποίηση τη οδηγία. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες Uh, να συμπεριλάβω τον εαυτό μου ε, στον κατάλογο των ομιλητών ως Ρηνιού. Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας, αλλά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπολογίζεται σε εμά του Ρηνιού, για την αναθεώρηση των προτύπων βάσει και της δουλειάς που γίνεται τώρα στον ΠΟΗ. Όπως είπατε, και το γράφετε και στο έγγραφο που έχουμε μπροστά μας, το να, στο, να θέσουμε τιμές οριακές είναι ένα μέρος της εργαλειοθήκης που θα πρέπει να φροντίσει να έχει η Ευρώπη θα πρέπει να γίνουν σεβαστά αυτά, διότι εάν δεν ορίσουμε τώρα τα όρια στο σωστό επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και τις προσπάθειές μας αναλόγως για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Το πρώτο σκέλος λοιπόν της στρατηγικής στα πλαίσια μιας πράσινης συμφωνίας είναι να ξαναδούμε ε, τις τιμές, τις οριακές τιμές, ε, μειωμένες, όχι αυξημένες, ε, και να κοιτάξουμε να προστατεύουμε καλύτερα την ατμόσφαιρα, τον αέρα που αναπνέουμε. Και μετά υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλο. Αφού ορίσουμε τι σωστέ τιμέ, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε κατανάλογα μέτρα που να συνοδεύουν την οδηγία πλαίσιο. Δηλαδή το ε, διοξείδιο του άνθρακα, η μείωση του άνθρακα, το να δουλέψουμε σε σχέση με τη χρήση φίλτρων σε κάποιε τεχνολογίε και ε, βιομηχανικού κλάδου. Θα έχουμε τι οριακέ τιμέ που θα ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα του ΠΟΕ και τι συστάσει του και μετά θα έχουμε και το ανάλογο νομοθετικό πακέτο, τη δέσμη μέτρων που θα επιτρέψει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Διότι ξέρουμε ότι προς στιγμή σήμερα δεν γίνονται σεβαστοί οι στόχοι. Και το νομοθετικό πακέτο αφορά κυρίως την ενέργεια, τις μεταφορές και την βιομηχανία. Και κάποιες φορές και τη γεωργία. Και σε συγκεκριμένε περιοχέ. Γι' αυτό περιμένουμε με ανυπομονησία τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι διαφορετικές στρατηγικές θα προτείνει. Την βιομηχανική πολιτική με μηδενικές εκπομπές, την κυκλική οικονομία και να κοιτάξουμε πώς επιτέλους θα γίνουν σεβαστά τα πρότυπα της ε, ατμοσφαιρικής ποιότητας που θα έπρεπε να ισχύουν ούτως ή άλλως. Ε, σταματώ εδώ και με την ιδιότητα του Προέδρου να δώσω το λόγο στους Πασίνους η κυρία Παύλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε ε, και ευχαριστώ που παρουσιάσατε τις διαφάνειές σας. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα, διότι αισθάνθηκα κάπως προδομένη. Για να δούμε πώς θα πάνε οι διαδικασίες στον ΠΟΗ και πώς θα ε, προχωρήσουμε δεν ξέρουμε ε, κατά πόσον η ισχύουσα οδηγία ε, εφαρμο... Ε, συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες του ΠΟΕ. Τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΗ σε κάθε περίπτωση. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί είναι γιατί να μην προχωρήσουμε λίγο γρηγορότερα και να προσαρμόσουμε κατευθείαν την οδηγία στα πρότυπα του ΠΟΕ. Αυτή είναι η πρώτη με ερώτηση. Και η δεύτερη Έχετε τίποτε μελέτες ή έρευνες για το θέμα που γίνεται όλο ένα και ε, πιο επίκαιρο για τα άκρος ε, λεπτά, τα μικροσκοπικά σωματίδια στη δική μου εκλογική περιφέρεια γίνονται έρευνες σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και έχει ε, βρεθεί ότι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε συγκεντρώσεις, υψηλέ συγκεντρώσεις ιδιαίτερα μικρών σωματιδίων έχουν μεγαλύτερη ε, τάση να αναπτύσσουν καρδιογειακέ παθήσεις και καρκίνο του κεφάλου. ID, ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινάω με ένα αστείο. Βάλτε τα ακουστικά σας. Σήμερα με το, ε, με το κορδόν σανιτέρ και τον αποκλεισμό ε, για υγειονομικούς λόγους περάσαμε μετά τους πράσινους σήμερα. Τέλος πάντων. Ε, για άλλη μια φορά χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για πραγματικούς λόγους υγείας όπως τον κορονοϊό που δημιουργεί τόσες ε, ανατεραχές αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Εσείς τέλος πάντων αναφερθήκατε ρητός σε μια πολιτική ομάδα Ήθελα λοιπόν να πω ότι εμένα αυτό που με απασχολεί είναι κάτι που απασχολεί και του άλλου συναδέλφου τη ομάδα ID που είναι και γιατροί. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον και η υγεία, ε, είναι ότι αυτό ε, το θέμα δεν μας απασχολεί εμάς λιγότερο από ότι άλλους συναδέλφους της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και όλων των άλλων. Οπότε καλό θα να αποφεύγετε τέτοιες, τέτοιους επενιγμούς. Ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να σας ζητήσω ένα σχολιασμό και ε, μια παρατήρηση για τη σημερινή συζήτηση για το κατά πόσο είναι κατάλληλη η οδηγία για την ατμοσφαίρη, κατάσταση της ατμόσφαιρας. Θα χρειαστούν ενδεχομένως αλλαγές σε σχέση λόγου χάρη με τους αποτεφρωτήρες, διότι περιμένοντας και επειδή έχουν περάσει, θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η κυκλική οικονομία και να μην έχουμε καθόλου απόβλητα, καταλαβαίνω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να θεωρεί ότι οι αποτεφρωτήρες είναι εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ώσπου να καταλήξουμε να έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία της κυκλικής οικονομίας. Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Η κυρία Χάζεκαμπ, από την ΓΚΟΕ, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω πως η ρήπανση η ατμοσφαιρική ρήπανση με τα λεπτά σωματίδια είναι πάρα πολύ βλαβερή για την αγία, για το περιβάλλον και για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, να σας πω πως οι εμπειρογνώμονες δεν συμφωνούν πάντοτε και δεν συμφωνούν με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει. Γι' αυτό είμαι ικανοποιημένη που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία ε, επί παραβάση κατά την κάτω χωρών και της Πορτογαλίας για αυτά τα σωματίδια τα οποία ορούνται σε πάρα πολλά σημεία και που πρέπει να σας πω βρίσκουν πολύ εύκολο το να περάσουν τα σύνορα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς έναν τόπο ασφαλή στην Ευρώπη. Ακόμα και πάρα πολύ μακρά από τις βιομηχανικές ζώνες, ξέρετε πως τα επίπεδα αυτών των σωματιδίων που αιρούνται είναι εξαιρετικά υψηλά και γι' αυτό εκ μέρους όλων των ε, πολιτών ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειωθούν οι εκπομπές αυτών των σωματιδίων, που είναι τόσο βλαβερές για την υγεία.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 We will now continue. Θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κινδύνους που έχουν να κάνουν, διατροφικούς κινδύνους με την εισαγωγή αλογίσιου κρέατος. Θα δώσω λοιπόν καταρχήν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Χάτσεν, έχετε το λόγο. Thank you very much, President. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω στην Επιτροπή σας για να εξηγήσω πώς έχει η κατάσταση. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί είμαι σίγουρος πως θα έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας κάποιες από τις βασικές παραμέτρους του θέματος αυτού. Καταρχήν, η βασική αρχή στην ευρωπαϊκή αγορά όλα τα τρόφιμα που διατίθονται στην αγορά, είτε είναι ευρωπαϊκής παραγωγής είτε εισαγόμενα, είναι ασφαλή και είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Ουσιαστική, θεμελιώδης αρχή, είτε είναι βόηο, είτε είναι χοιρινό, είτε είναι αυγά, είτε είναι αλογίσιο κρέας. Τώρα, για το κρέας αλόγου, εδώ είναι μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο προϊόν. Είμαστε η βασική αγορά, είμαστε μία από τις λίγες περιοχές του κόσμου που είναι ε, βρόσιμα τα άλογα και σε επίπεδο εισαγωγών εισάγουμε αλογίσιο κρέας από τρίτες χώρες όπου ε, συμμορφώνονται με μια σειρά από προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα η τρίτη χώρα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη η τρίτη χώρα. Οπότε έχουμε επαληθεύσει πως έχουν καλές κτηνιατρικές υπηρεσίες με τις απαραίτητες δομές. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο εγκεκριμένο ε, παρακολούθησης ε, καταλήπων και υπολοιμάτων. Και τρίτον, ε, ένας κατάλογος συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Γιατί το τονίζω, γιατί ε, λειτουργούν σωρευτικά. Αν εξασφαλίζεις μόνο το ένα ή δύο από αυτά, δεν έχεις δικαίωμα να ε, κάνεις εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλες, όλες οι παρτίδες θα πρέπει να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό και γίνονται οι συνηθισμένοι έλεγχοι πάντοτε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις εμπορίου με τρίτη χώρα, οι επιθεωρητές μας τακτικά κάνουν επισκέψεις για να επαληθεύσουν πως οι χώρες αυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσει τις οποίες ε, μόλις παρουσίασα και τις οποίες έχουμε θέσει και όπου προκύπτουν ζητήματα κάνουμε follow-up με τις χώρες αυτές και ξέρετε κι εσείς πως στο παρελθόν είχαμε πολύ αυστηρή δράση για παράδειγμα με τη Βραζιλία όταν είχαμε βασικές ελλείψεις οι οποίες ανακαλύφθηκαν. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή πέντε μόνο χώρες παγκοσμίως είναι εγκεκριμένες για να εξάγουν αλλαγή κρέα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργεντινή, Αυστραλία, Καναδάς, Ελβετία και Ουρουγουάη. Και πρέπει να πω εδώ πως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του εμπορίου προέρχεται από την Αργεντινή και δεύτερο, ε, δεύτερη μετά την Αργεντινή, σε εξαγωγές είναι η Ουρουάη. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο και θα μπορούσα τώρα να ακούσω τις ερωτήσεις σας και με μεγάλη χαρά θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χάτσον για τα σχόλια αυτά. Είμαι η πρώτη που θα ξεκινήσει με αυτά που έχω να πω, γιατί εγώ ε, υπέβαλα το αίτημα να έρθετε και θα το κάνω στα Ολλανδικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει χιλιάδε τόνου ε, αλογίσου κρέατο από την Αργεντινή και τον, την Ουρουάη. Από το 2011 ειδοποιούν οι περιβαλλοντικέ με κυβερνητικέ οργανώσει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ζωική υγεία και ευζοία ω προ τα θέματα αυτά. Και το Ίδρυμα για την Ευζοία των Ζώων λέει ότι έχει παρακολουθήσει την κατάσταση στην Νότια Αμερική, ιδίως το 2019, και σε αυτήν την διεξοδικότατη έκθεση έχουν καταλήξει ότι τα άλογα εγκαταλείπονται στην τύχη τους επί εβδομάδες ε, χωρίς, ε, σε ειδικά κέντρα χωρίς ε, τροφή, χωρίς νερό, χωρίς έλεγχο της υγείας τους. Τα άλογα αυτά δεν έχουν καμία φροντίδα και τα αφήνουν εκεί να πεθάνουν πολλές φορές με ηλεκτροσόκ. Κανένα από τα πρότυπα για την ευζοία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τηρηθεί. Πολλέ φορέ έχουν λάβει βαριά φάρμακα και καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα ενώ του αλλάζουν απλώ τις ετικέτε. Το 2018 η Γενική Διεύθυνση Σάντα έχει λάβει γνώση και υποτίθεται ότι έγιναν έλεγχοι, οι οποίοι όμως σαμποταρίστηκαν όταν έφτασαν επιθεωρητές για να κάνουν τους ελέγχου του, Ξαφνικά δεν υπήρχαν ε, ζώα στα σφαγεία ή στα κέντρα ε, συγκέντρωση των αλόγων. Αν διαβάσω λοιπόν προσεκτικά την έκθεση των Ευρωπαίων Επιθεωρητών, λέει ότι κατά τι τέσσερι ημέρε η αποστολή παρακολούθηση ε, διαπίστωσε ότι ήταν εντελώ ακατάλληλε οι υποδομέ για τον αριθμό των ελόγων που αναφέρονταν στην έγγραφα. Επιπλέον, ε, υπήρχαν ε, κακές, ήταν κακή κατάσταση των στεγών και οι υγειονομικέ συνθήκε στα κέντρα συλλογή δεν διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι συστάσεις και τα πρότυπα των διεθνών οργανισμών. Δεν υπήρχαν βέβαια εκεί ζώα, ούτε στα κέντρα ούτε στα σφαγεία, όμως οι υπεύθυνοι έλεγαν ότι όταν λειτουργούν ε, τα κέντρα, σίγουρα η υγεία των ζώων θα βρισκόταν υπό απειλή. Η αρμόδια αρχή λοιπόν δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι οι αρχές που, που διέπουν την ε, κοινή αγορά ε, και οι επιταχές για την δημόσια υγεία τηρούνται. Επίσης, τα ιατρικά και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται στα άλογα δεν χορηγούνται βάσει των ετικετών των οδηγιών χρήσης ή των ημερομηνιών λήξης. Η υγεία λοιπόν των ζώων ε, είναι κάτι που το έχουν ε, επισημάνει ως πρόβλημα στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη και οι αρχές της Επιτροπής που έκαναν οι ίδιες τον έλεγχο, αλλά και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πώς γίνεται λοιπόν δύο χρόνια αργότερα να συνεχίζει να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλογίσιο κρέα από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη, θα έπρεπε με όσα έχουν διαπιστωθεί να έχει απαγορευτεί η εισαγωγή οποιοδήποτε κρέατο από τι χώρε αυτή. Ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται τα πορίσματα των αποστολών. Ε, η Επιτροπή λέει ότι με τη συνθήκη Μερκοσούρ θα σταματήσουν να επιβάλλονται δασμοί σε αυτό το είδου το αλογίσιο κρέα στο μέλλον. Ακόμα λοιπόν λιγότερη έλεγχη για την ασφάλεια αυτών των ε, ζωντανών Πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δικαιολογήσει τη μείωση των ελέγχων για αυτό το είδος το κρέας, ενώ όλα δείχνουν ότι δεν είναι ασφαλές. Είναι λογικό να συνάψουμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών αυτές τις χώρες υπό το φω αυτών των ε, αποκαλύψεων. Εγώ πιστεύω πως όχι. Η κυρία Νέτ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στην τελευταία τη επιθεώρηση για το αλλαγή κρέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα και υπόθηκε ήδη ότι η ευζοία των ζώων και οι κανόνε ασφάλεια των τροφίμων δεν τηρούνται. Η έκθεση αυτή παραδέχεται ότι δεν μπορούμε να θυσιάζουμε τις απαιτήσει της δημόσιας υγείας της ευρωπαϊκής αγοράς για τις εισαγωγές. Εμείς ε, κάνουμε ελέγχους για τα κτηνιατρικά προϊόντα και για λόγους ίχνη λασιμότητας και προέλευσης των αλόγων ε, βλέπουμε στην άλλη πλευρά, στην Νότια Αμερική, να επικρατεί ένα μυστήριο. Εδώ και χρόνια τα πορίσματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων αυτό δείχνουν ότι ισχύει και για την Αργεντινή και όχι μόνο για την Ουρουάη. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε τις εισαγωγές προϊόντων που ξεκάθαρα δεν σέβονται τα πρότυπα ευζοίας των ζώων. Πρότυπα που τουλάχιστον να είναι κοντινά στα δικά μας. Θα αποφύγω να σας αναφέρω όλα αυτά τα δυσάρεστα και στενά χωρά που συμβαίνουν στα κέντρα συγκέντρωση όπως λέγονται και στα σφαγεία. Ένα απλό παράδειγμα, κανόνες μεταφοράς των αλόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 24 ώρες και κάθε 8 ώρες διακοπή για φαΐ και νερό. Στην Αργεντινή 36 ώρες χωρίς νερό ούτε τροφή. Στην Ουρουγουάη δεν υπάρχουν καν κανόνες. Αυτά ε, παραμένουν απάνθρωποι, σκληρή μεταχείριση ε, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων και ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να ξεκουνηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ερώτηση τη δική σας και της ε, συναδέλφου σας. Καταρχάς, χαίρομαι που διαβάζετε τις εκθέσει των κτηνιατρικών μας υπηρεσιών με τέτοια προσοχή. Όχι σοβαρά το λέω. Είναι σοβαρό. Διότι πραγματικά δαπανούμε τεράστιες προσπάθειες, χρόνο και δουλειά για να γίνουν όλα αυτά και ακριβώς έτσι μπορούμε να έχουμε πακριβή γνώση του τι συμβαίνει στην πράξη. Για να στραφώ στην ε, κατάσταση και τις διαφορές που αναφέρατε θέσατε, γύρατε ερωτήματα για την Ουρουάη και την Αργεντινή. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις λοιπόν πρώτα. Καταρχάς, και νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί ξανά στην Επιτροπή σας, επανειλημμένος ε, στο πέρας των ετών. Σε ό,τι αφορά την ευζοία των ζώων, τα πρότυπα που μπορούμε να επιβάλλουμε σε εμπορικούς μας εταίρους είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τα σφαγεία μόνον την ε, στάση και, την, ε, και τα σφαγεία. Δεν έχουμε την αρμοδιότητα να επιβάλλουμε ευρωπαϊκούς κανόνες σε γενικότερα θέματα ευζωίας. Ε, υπό το φως αυτής της παρατήρησης αναμένουμε οι εμπορικοί μας εταίροι να σέβονται και μια σειρά από άλλους κανόνες ό,τι αφορά τη διοργάνωση των σφαγείων και ούτω καθεξής μια σειρά από στοιχεία και στην τελευταία έκθεση για την Ουρουγουάη και την Αργεντινή ε, δείχνουν ότι υπάρχουν ελλείψεις. Και το κοιτάμε το θέμα. Σε ό,τι αφορά την Αργεντινή, να σας ενημερώσω ότι η συνολική μας αξιολόγηση για τις απαντήσεις που λάβαμε από τις αρμόδιες αρχές της Αργεντινής επί χάρτου φαίνονται καλέ. Μπορεί να πείτε βέβαιος ότι επί χάρτου και σε ένα έγγραφο όλα καλά ακούγονται. Αλλά πραγματικά η ομάδα μα, ε, η ομάδα επιθεωρητών μα, πρόκειται να προσγειωθεί όπου να είναι ή μόλι έχει προσγειωθεί στην Αργεντινή για να κάνει ένα δεύτερο γύρο ελέγχων. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε σε σχέση με του εταίρου μα. Μόλι δούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κοιτάζουμε να πάρουμε ικανοποιητική απάντηση από τι αρμόδιε αρχέ, όπω κάνουν τα κάτι μέλη, και μετά όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, πάμε και κοιτάζουμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο ελέγχων. Όπως είπα, ε, στην περίπτωση της Αργεντινής πιστεύουμε ότι στο χαρτί τα πράγματα δείχνουν ότι ασχολούνται να βρουν λύσεις στα βασικότερα προβλήματα. Τώρα για την Ουρουγουάη δεν έχει γίνει τέτοια πρόοδος. Συζητάμε ακόμα μαζί του και έχουμε ε, την ελπίδα ότι σύντομα θα γίνει και δεύτερος γύρος ελέγχων και εκεί. Σε ό,τι αφορά την συμφωνία Μερκοσούρ και τι θα προκαλούσε ή όχι. Είχα την ευκαιρία πριν από τα Χριστούγεννα σε μια άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου να εκθέσω το τι θα συνέβαινε σε σχέση με τα θέματα φυτογενομικής και κτηνατικής υγείας. Εδώ το βασικό είναι ότι τα προϊόντα θα πρέπει να φτάνουν στο ύψος των προτύπων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εισάγονται στην ε, Ένωση τα, οι έλεγχοι θα παραμείνουν. Ωστόσο, αυτό που θα παραμείνει σίγουρα είναι μια ε, διάταξη, ρήτρα, για να έχουμε διάλογο γύρω συζητήσεων για θέματα ζωή, ε, των ζώων. Διότι συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε που εκφράσατε εδώ σήμερα το απόγευμα. Και μπορώ να σα βεβαιώσω ότι έχουμε εργαστεί αόκνο με τι ε, χώρε εταίρου για να προσπαθήσουμε να ε, του πείσουμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσληψη των προτύπων. Ε, και θέλω να σα διαβεβαιώσω, κυρία Χάζεκαμπ, η προσοχή που δίνουμε στην ευζοία των ζώων παγκοσμίω είναι πολύ μεγάλη στην Ευρώπη. Είμαστε βεβαίω πρωτοπόροι, αλλά προσπαθούμε να προωθήσουμε τα πρότυπά μα και στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι οι κανόνε πέραν των σφαγίων δεν μπορούν να επιβληθούν με άλλο τρόπο, διότι είναι εκτό του πλαισίου υγιεινή και φυτογενή ε, Πάντω σα διαβεβαιώ ότι τα θέματα αυτά πραγματικά τα παρακολουθούμε, τα κοιτάζουμε με προσοχή και βεβαίω εφόσον το επιθυμείτε είμαστε στη διάθεσή σα να σα ξαναενημερώσουμε όποτε το επιθυμείτε είναι αυτό το χρόνο. Ελπίζω ότι απήντησα στα ερωτήματα που τέθηκαν τουλάχιστον σε γενικέ γραμμέ. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει σα. Βεβαίω θα φροντίσουμε να σα ξαναενοχλήσουμε μόλι ολοκληρωθεί ο δεύτερο γύρο ελέγχων και. Ε, Ελπίζουμε να μην καταλήξουμε και πάλι στα ίδια συμπεράσματα με βάση των νέων πορισμάτων που θα έχετε ως τότε. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της συνεδρίασης. Αύριο η συνεδρίασή μας θα συνεχιστεί στις 11 με ανταλλαγή απόψεων με, τον, με την κυρία Κυριακίδη, την Ευρωπαία Επίτροπο.